δάσετε στη μονομερή επαναφορά των απαιτήσεων ε, θεωρήσεων από τον Καναδά για τους Τσέχους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει το, ε, το Συμβούλιο να λάβει μέτρα όσον αφορά ε, το Καναδά, ούτω ώστε να καταργηθεί αυτή η απέτηση για θεώρηση ταξιδίων, θεώρηση διαβατηρίων για τους Τσέχους υπηκόους. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους πολίτες της τσεχικής δημοκρατίας που όπως οι άλλοι ε, υπήκοοι των ε, κρατών των άλλων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έπρεπε να μπορούν